μας, την πλήρη μας Σας καλωσορίζουμε πάντως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα θα ψηφίσουμε και πρώτα απ' όλα πρώτα απ' όλα λέγω Α, η κυρία Ροντσέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από Λίγα δευτερόλεπτα είναι αυτά για να εκφράσω τη διαφωνία μου όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου να απορρίψει την έκθεση ε, στρέλο όσον αφορά τη γονική άδεια. Σήμερα εκφράζω διάφορες μητέρες και πατέρες της Ευρώπης που απογοητεύτηκαν πάρα πολύ από την απόφαση του Συμβουλίου. Είναι μια έλλειψη υποστήριξη των αξιών και καταδικάζω αυτό, μόνο μου το είναι. Προ ποια Ευρώπη κινούμαστε. Το να απορρίπτονται προτάσει ήταν μια επιλογή που στρέφεται κατά των οικογενειών του σήμερα, αλλά κυρίω κατά των οικογενειών του αύριο. Ευχαριστούμε κύριε Ροντσέλη. Τώρα θα ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Μπέργκε. για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις πλημμύρες στην Πορτογαλία και τις ε, θεομηνίες στη Γαλλία. Είναι ονομαστική η ψηφοφορία με ενισχυμένη πλειοψηφία. Ενισχυμένη. Έληξε. εγκρίνεται. Τώρα η έκθεση Σουριάν για το, για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού είναι ονομαστική επίσης ψηφοφορία άρχεται. Έληξε. έληξε είπα και αυτό εγκρίνεται. Τώρα η έκθεση της κυρίας Ματέρα για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής προς την Παγκοσμιοποίηση. Η πρώτα για τη Σλοβενία. Είναι και αυτή η ενιαία και ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται με ενισχυμένη πάντα πλειοψηφία. Έληξε. Εγκρίνεται για το ίδιο θέμα, αλλά αυτή τη φορά για την Χαϊδελβέργη, πάλι ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται ίδιο θέμα αλλά για την πολωνική αυτοκινητοβιομηχανία ονομαστική άρχεται. Και πάντα απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία. Έληξε. Εγκρίνεται. Ίδιο θέμα αλλά για το ισπανικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο άρχεται η ψηφοφορία, πάλι τα ίδια δηλαδή, ονομαστική και ενισχυμένη. Έληξε. Εγκρίνεται. Το ίδιο θέμα αλλά για την υφαντουργία στη Βαλένθια άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. Το ίδιο θέμα αλλά αυτή τη φορά για την φυσική πέτρα. Στη Βαλένθια πάλι. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται πάλι το ίδιο θέμα αλλά αυτήν τη φορά για το ΛΕΑΡ στην Ισπανία ονομαστική ψηφοφορία άρχεται έληξε εγκρίνεται το ίδιο θέμα αλλά για το Πόσναν στην Πολωνία ονομαστική ψηφοφορία άρχεται έληξε εγκρίνεται ευχαριστούμε την κυρία Ματέρα είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για αυτή την κινητοποίηση είναι σήμερα ικανοποιημένοι τώρα η έκθεση του κυρίου Μωράς για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003 109 κάθετος CE Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Τώρα η έκθεση της κυρίας Γκρισμπέκ για μια συμφωνία ένωσης και γεωργίας για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Α, όχι, δεν είναι ονομαστική, δεν είναι ονομαστική. Διάρσεως της χειρός. Είχα συνηθίσει να λέω ονομαστική και το είπα και αυτή τη φορά λοιπόν. Έκθεση Γκρίσμπεκ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Τσανίκη για μια γρήγορη ανταπόκριση. Ονομαστική ψηφοφορία αυτή τη φορά άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Η έκθεση τώρα της κυρίας Σουίνμπουρν για ορισμένα δημοσιονομικά εργαλεία, dark pools και τέτοια. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Γκόμες για την ενίσχυση της ασφάλειας στον χημικό, βιολογικό και άλλους τομείς. Η εισηγήτρια έχει ζητήσει το λόγο. Και τα ραδιολογικά, τα πυρηνικά υλικά ε, δεν, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Δημιουργούν φυσικές καταστροφές. Αν υπάρξουν ποινικέ καταστροφέ, οι καταστροφέ δεν γνωρίζουν σύνορα. Έχουν καταστροφικέ συνέπειε στην ανθρώπινη ζωή για τι υποδομέ, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Όταν συμβαίνουν καταστροφέ αυτού του είδου δεν γίνονται κάπου μακριά. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ουγγαρία ε, σχετικά πρόσφατα. Και μετά τα πακέτα μετακριτικά που απεστάλησαν προς διαφόρους ε, προορισμούς από την Ιεμένη, προς τη ΣΥΠΑ και τις χώρες της Ευρώπης. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να βελτιωθεί η συνεργασία που απαιτείται όσον αφορά το δυναμικό που έχουν τα κράτη-μέλη για να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν τέτοιου επιθέσεις. Χρειάζεται ειδικό μηχανισμό Ευρωπαϊκό για να βρίσκονται απαντήσεις σε αυτού του είδους κρίσεις. Καθώς χρειάζεται και συνεργασία σε θέματα συνεργασίας των δυνάμεων αστικής προστασίας. Χρειάζεται ενίσχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά που ενέκρινε το Συμβούλιο του 2009 δεν αρκούν. Ένα πρόγραμμα που δεν εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη. θα πρέπει, αν σπάσει μια λυσίδα, με ένα κρίκο αλυσίδα, καταραίει όλη η αλυσίδα. Άρα χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων τα κάτι μέλη. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία στον πολιτικό και στεντικό τομέα και συντονισμό των προσπαθειών όσον αφορά την πρόληψη, προστασία και απάντηση όταν συμβαίνουν διάφορε τέτοιε καταστροφέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα συστήματα προστασία. Το σχέδιο δράση για την ασφάλεια κατά χημικών, ραδιολογικών, πυρηνικών ε, τέτοιων ε, συμβάντων ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα αυτά που προβλέπει η συνθήκη τη Ευχαριστώ κυρία Γκόμε για αυτή την εξήγηση. Πάμε στην ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εκθέση για την καλή διακυβέρνηση, την έκθεση Μανέσκου. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Και πάμε στην έκθεση Δίας μέρα όσον αφορά τη δημιουργία ε, ενός δικτύου ε, αρμοδίων για θέματα μετανάστευσης. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ας ψηφίσουμε την τροποποιηθήσα πρόταση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και ονομαστική ψηφοφορία για να ψηφίσουμε το ψήφισμα αναφορετικού περιεχομένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και η έκθεση εγκρίνεται. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση Ματιού Υπάρχουμε τεράστιο, πολύ μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Λοιπόν, σας παρακαλώ να σηκώνετε καλά το χέρι σας, μην κουραστείτε στα μισά του δρόμου και σταματήστε να σηκώνετε το χέρι σας. Παρακαλώ να είσαστε σε φόρμα, να κατευθείτε σε φόρμα, θόλη τη διάρκεια τη ψηφοφορία. Σηκώντε ψηλά το χέρι, αλλιώ τελικά θα καθυστερήσουμε. Α ψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση Ματιέ όσον αφορά τη διαδικασία ενιαία αίτηση για άδεια παραμονή και εργασία. Έχουμε 36 τροπολογίες που ψηφίζονται μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τώρα προχωράμε και πάμε σε μια ομάδα τροπολογιών της Επιτροπής της Αρμόδιας, η τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο. Ας κάνουμε έλεγχο για τη 13. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 16, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Οπότε τώρα ψηφίσουμε την τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές θα γίνει έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 18. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στη 19, τροπολογία 19. Υπέρ. Ας δούμε τα χέρια να σηκώνονται κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν τα βγάζουμε πέρα έτσι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι μικρές οι διαφορές, 6-7 ψήφοι διαφορά, γι' αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορία. σαφής η διαφορά, εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Ας δούμε τα χέρια. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εντάξει. Α κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 51. Ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται σαφώς. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 65 ονομαστική ψηφοφορία ξεκινάει Τέλος ψηφοφορίας. Σαφώς εγκρίνεται. Η επόμενη τροπολογία είναι 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74 τώρα. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 73. Ξεκινάει. Τροπολογία 73. Τέλος. Απορρίπτεται. 73 υπέρ, 74 συγγνώμη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ας προχωρήσουμε και πάμε στην 89 υπέρ, κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε έναν έλεγχο. Ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα να ψηφίσουμε την 90. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 30 απερίφθη. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 91. Ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. 91. Πέρας εγκρίνεται. Η επόμενη είναι η 119 ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Οπότε θα ψηφίσουμε τώρα την 31, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. 31. Πέρας. γκρίνεται Και αυτό σημαίνει ότι 113 καταπίπτει. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε την 120, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 32. Ονομαστική ψηφοφορία και πάλι ξεκινάει για την 32. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 114 συνεπώς καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 34 με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τροπολογία 34. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Και καταπίπτει η 115. Ψηφίζουμε τώρα δύο ταυτόσιμες τροπολογίε στην 36-121, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καταπίπτει η 43. Περνάμε στην 93 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ. 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 93. 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, υπέρ, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται από ό,τι φαίνεται. Ε, εγκρίνεται η 94. 95 παρακαλώ, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έτσι καταπίπτει η 48. Τώρα η 50 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 96 υπέρ κατά άποχες. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ, νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Επαληθεύουμε. ονομα ε, Ψηφοφορία για την 96. Πέρας. Όντως απερίφθη. 97 υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. 97. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 54. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 95, 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά ας την επαληθεύσουμε. 99 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της προφορίες. Εγκρίνεται 99. Πολύ καλά. Υπαριθμών 100 τροπολογία υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 57. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές έχει εγκριθεί μάλλον, αλλά ας δούμε. Η 101 παρακαλώ, επαλήθευση. Πέρας της προφορίας. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κύριε Σπερώνη, ζητάτε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορούμε τον κατάλογο των τροπολογιών στον πίνακα να τον ανανεώσουμε. Παρακαλώ. Στην οθόνη. Ναι, Πρόεδρε, το εξετάζουμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σπερόνι, το εξετάζουμε. Αλλά εσείς το βλέπετε στη δική σας την οθόνη, έτσι δεν είναι. Ας προχωρήσουμε. 103. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 103 εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 67. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 107. Πέρας. Εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Καταπίπτει η 68. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται η 111, καταπίπτει 69 και ψηφίζουμε την 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι πρόεδροι ομάδων παρακαλώ να σηκώνουν και εκείνη το χέρι γιατί δεν τους βλέπω. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 77 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 77 και έτσι καταπίπτει η 116 στην 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και έτσι ψηφίζουμε την 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα μαζί την 11 και την 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, εγκρίνονται, εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε τη 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και έτσι ψηφίζουμε την 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε την 82. Επαληθεύουμε για την 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται όντως. 117 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Έτσι ψηφίζουμε την 83 πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η 83. Και έτσι ψηφίζουμε την 118 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίψετε 118. 84. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 86 καταπίπτει η 14. 87 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η 87. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και η 88. Τώρα το σύνολο της προτάσεως όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης επιτροπής όπως τροποποιήθηκε υπέρ ε, άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται se nota, ¿no? ¿Sí? Vale, vale, vale, vale. Bueno, dado que, dado que la propuesta... Δεδομένου ότι απερίφθη η πρόταση, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. La señora comisaria, Κυρία Επίτροπε, διορθώνει ο Πρόεδρος. Um, Κύριε Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ότι εγώ απλώς ακούω, παρακολουθώ και έλαβα το μήνυμα που μας δώσατε. Είναι σαφές. Σας υπόσχομαι. Θα το μεταφέρω, θα το μεταφέρω. Αντικειμενικά, διότι είδα τι έγινε. Οι συνάδελφοι θα επανέλθουν αφού το ξανασυζητήσουν στο σώμα των Επιτρόπων. Καλά. Τώρα επανυποβάλλεται στην Κομισιόν η πρόταση αναπέμπεται. Και τώρα η έκθεση... Α, τι θέλετε κύριε Φερκές. Τι θέλετε κύριε Φερκές. Κύριε Πρόεδρε, με βάση τα άρθρα 175 και 6 θέλουμε να μάθουμε αν η Κομισιόν θα αναθεωρήσει την πρόταση αυτή και θα την επανυποβάλει γιατί δεν είναι αυτόματο κάτι τέτοιο. Πρέπει να μας πει τώρα αν αποσύρει την πρόταση ή αν θα την επανυποβάλει στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, άκουσα αυτά που είπε η κυρία Επίτροπος και συνεπέρανα ότι θα επανυποβάλει, αλλά θα τη ρωτήσουμε και ρητά να μας πει ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Ορίστε κυρία μου, σας παρακαλώ πέστε μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούστε. Με εκπλήσει αρκετά το ότι βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση ε, και συνδιαλλαγή εδώ και ένα χρόνο. Είχαμε επιτύχει συμφωνία με τους φιλελεύθερους και βλέπω την τελευταία στιγμή ότι ψήφισαν διαφορετικά αντίθετα από τη συμφωνία που είχαμε συνάψει. Διαπιστώνω ότι η συμφωνία μου λέω με τους φιλελεύθερους δεν έχει τηρηθεί ενώ είχαμε φτάσει στην Ολομέλεια με άλλες συμφωνίες και ο κύριος Σαρκάς προτείνει κοιτάξτε αφήστε με να τα πω λοιπόν οι σοσιαλιστές προτείνουν η Κομισιόν οι σοσιαλιστές και ιδιαίτερα ο κύριος Σαρκάς προτείνουν η Κομισιόν να αναπέμψει την πρότασή της Ακούστε όμως κύριε Σαρκάμου, εδώ και ένα χρόνο το συζητάμε. Και εδώ και ένα χρόνο προτείνεται πράγματα που απορρίπτονται. Τι νόημα έχει λοιπόν να ξαναρχίσουν όλα αυτά και δέκα χρόνια να τα πούμε ποτέ δεν θα συμφωνήσετε Αλέξανδρε. Κάναμε όλες τις προσπάθειες που μπορούσαμε να κάνουμε και ποτέ δεν συμφωνούσατε. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω με τι τρόπο άμα συνεχίζετε απλώς να κάνετε τις ίδιες προτάσεις θα προχωρήσουμε. Κρίμα, πολύ κρίμα. Είχαμε πει όλοι όσοι μεταναστεύουν εδώ να έχουν ίση μεταχείριση το αρεπορρίπτουν αυτό οι σοσιαλιστές την εξίσωση της μεταχείρισής τους με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους ενώ είχε συμφωνηθεί κάτι τέτοιο σας παρακαλώ, λέει ο πρόεδρο, σα παρακαλώ αφήστε τα ου. Δεν θέλω ου. Αφήστε λέγω τα ου για να εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Η Κομισιόν πρέπει να μας πει αν θα διατηρήσει την πρόταση αυτή αναθεωρημένη ή όχι. Αφήστε λοιπόν την κυρία Επίτροπο να μας το πει. Είπε ότι θα μεταφέρει αντικειμενικά το μήνυμα, εντάξει, αλλά να μας πει επίσης και αν διατηρεί την πρότασή της ή όχι. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε αν μετά από αυτήν τη συζήτηση που είχε τόσο πάθος βγάλω το συμπέρασμα ότι στις Βρυξέλλες θα συνεδριάσει το Κολέγιο των Επιτρόπων και θα δούμε τι θα αποφασίσει αφού συζητήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Άρα λέει ο πρόεδρος η κυρία Επίτροπος μόλις μας είπε ρητά το εξής ότι προς στιγμήν δεν αποσύρει την πρότασή της αυτό μας είπε και μετά θα δούμε τι θα γίνει Λοιπόν, η Κομισιόν δεν αποσύρει λοιπόν την πρότασή της, μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στην έκθεση της κυρίας Χιμένες Μπεσερίλ και της κυρίας Ρομέρο για την ε, απόφαση ευρωπαϊκής προστασίας. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για να δούμε τώρα. Να δούμε λοιπόν. Θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου. Μα εδώ ψηφίζουμε κυρία Χιμένες Μπεσεριλ. Τι θέλετε. Ορίστε, ορίστε. ορίστε. Ζήτησα το λόγο για να σας υπενθυμίσω τη σημασία της σημερινής ψηφοφορίας για να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο ως προς τις χώρες που δεν έχουν ακόμη λάβει αυτά τα μέτρα προστασίας. Εδώ θέλουμε την προστασία των θυμάτων για να μπορέσουν να διαβιώσουν, να ζήσουν χωρίς τον φόβο. Τα παιδιά, οι γυναίκες που είναι θύματα τρομοκρατίας, το εμπόριο, λευκής σαρκός κτλ. Α, κάλλιστα λέει ο Πρόεδρος. Α, και η κυρία Ρομέρο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέμα αυτό θα ήθελα να επινθύσω στους φιλελεύθερους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί αυτό το κείμενο για την πράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και άλλες κυβερνήσεις ακόμα δεν έχουν προσυπογράψει αυτό το σχέδιο και θα ήθελα να δω αν θα υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Αφού ακούσαμε τους δύο συγγητές ε, και αφού εγκρίναμε την τροπολογία θα ψηφίσουμε την τροποποιηθή σε πρόταση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματο του θετικού περιεχομένου με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. Εγκρίνεται. Με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια λοιπόν στους ηγητές. Προχωράμε και πάμε στην έκθεση της κυρίας Μπάουερ και κυρίας Χέντ για την εμπορία ανθρώπων. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε το πρωτότυπο κείμενο. Το άρθρο 2 παράγραφος 1. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Πέρας. Εγκρίνατε. Τροπολογία 3 υπέρ. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα πάμε για να ψηφίσουμε την πρόταση που τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και το σχέδιο ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μια συντριπτική πλειοψηφία και ψηφίζουμε την έκθεση Γκρίσμπεκ τώρα όσον αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν ε, άνευ Δεν υπάρχουν τροπολογίες, οπότε θα ψηφίσουμε κατευθείαν το σχέδιο ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα έκθεση Λούχαν για εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Παράγραφος 6, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Τέρας, πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ο κ. Μελό. vale, vale. Sí, sí, yo te he visto. Te he visto, te he visto. Le bot, de materia de tu. A las explicaciones de voto. Εξηγήσεις ψήφου. Πρώτος, όσον αφορά την έκθεση Μωρές ο κύριος Μαστέλα. Τέλα νοστά.